Ακολουθεί η δήλωση της υπάτης εκπροσώπου της Ένωσης για τις εξωτερικές υποθέσεις και την πολιτική ασφαλείας διπροέδρου της Επιτροπής κυρίας Άστον με θέμα τον σεισμό στην Αιτή. Θα λάβει το λόγο επίσης ο Επίτροπος Ντεχόχτ στη συνέχεια, αλλά πρώτα η κυρία Κάθριν Άστον και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω την ευκαιρία την καλωσορίσω μετά από τη μακρά συνεργασία που είχαμε σε άλλου τομεί και της εύχομαι κάθε επιτυχία κατά τη διάρκεια των καθηκόντων σα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο, δηλαδή, Άστον. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Θα μου επιτρέψετε να σας ενημερώσω για την κατάσταση στην Αϊτή μετά από την φρικτή τραγωδία της 12ης Ιανουαρίου. Οι απώλειες είναι τεράστιες, όπως και οι ζημίες. Τρία εκατομμύρια κόσμος έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την τραγωδία αυτή και ο αριθμός των ε, νεκρών αυξάνεται. Πρόκειται επίσης για μια ανθρωπιστική καταστροφή, για μια πολιτική καταστροφή και συνεργαζόμεθα με τα Ηνωμένα Έθνη και με την ηγεσία την Αιτινή για να προσπαθήσουμε να ελαφρύνουμε τον πόνο τους. Το θέμα είναι να βοηθήσουμε την IT μακροπρόθεσμα και αρκετοί πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν χάσει τη ζωή τους και αγνοούνται περίπου χίλιοι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς αντιδράσαμε γρήγορα, δεν επιζητήσαμε τα πρωτοσέλιδα αλλά απευθεία στείλαμε βοήθεια. Μετά από τη γνώμη των Ηνωμένων Εθνών δεν ταξιδέψαμε αμέσως στην Ταϊτή, κάτι το οποίο θα προκαλούσε πάρα πολλά έξοδα και θα απομάκρυνε την προσοχή από το πραγματικό πρόβλημα. Συμφώνησα λοιπόν και με τον Επίτροπο Ντεγκούχτ, ο οποίο θα μεταβεί στην ΑΕΤ αυτή την εβδομάδα για να μεταφέρει τα συλληπιτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να επαναλάβει την αφοσίωσή μας στην προσπάθεια ανοικοδόμησης θα συζητήσει τη βοήθεια που έχει δοθεί μέχρι τώρα και θα συζητήσει επίσης με τα Ηνωμένα Έθνη τις πιο πιεστικές ανάγκες της χώρας για τους επόμενους μήνες. Εν Συνεχίζουμε να προσπαθούμε με κάθε τρόπο και στον ανθρωπιστικό τομέα και στον πολιτικό τομέα και στον τομέα της ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών ήμουν σε συνεχή επαφή με την Υπουργό Κλίντον, με τον Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, με Υπουργούς Εξωτερικών διαφόρων χωρών, μεταξύ των οποίων και του Καναδά, ο οποίος ηγείται της ομάδας φίλων χωρών της ΑΙΤΙΣ. Προσπαθούμε να συντονίσουμε την διεθνή ανταπόκριση. Θα ταξιδέψω αυτή την εβδομάδα στις Ηνωμένε Πολιτείε για να συζητήσω τα θέματα αυτά με την Αμερικανική κυβέρνηση και τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και άλλους στη Νέα Υόρκη. Τα Ηνωμένα Έθνη ζήτησαν κατεπίγουσα οικονομική βοήθεια άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων όπως και επιμελητιακή βοήθεια για τη μεταφορά της βοήθειας. Χθες ο Γενικός Γραμματέας Μπαν ζήτησε επίσης ενισχύσεις ε, για την δύναμη των Ηνωμένων Εθνών για την τήρηση της τάξης. Ζήτησα επίσης και από την Ισπανική Προεδρία να συγκαλέσει χτες ένα έκτακτο συνέδριο, ε, συμβούλιο μάλλον υπουργών εξωτερικών, για να συντονίσουμε σωστά και τις προσπάθειες της Γραμματείας του Συμβουλίου, των κρατών μελών και της Επιτροπής έτσι ώστε με ένα ολοκληρωμένο τρόπο υπό την κατεύθυνσή μου να προσπαθήσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Αυτό είναι μια καινοτομία. Χθε ήταν θα έλεγα παραγωγική συνάντηση που έγινε και όλοι θελήσαμε να ενισχυθεί η συνεργασία μας με τα Ηνωμένα Έθνη σε επίπεδο οικονομικής βοήθειας. Καταλήξαμε στα εξή άμεση ανθρωπιστική βοήθεια από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή 30 εκατομμυρίων δολαρίων. 92 εκατομμύρια σε συγκεκριμένες πιστώσεις υποχρεώσεων από πλευρά των κρατών μελών. Αυτό θα καλύψουμε τα 100 εκατομμύρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μη ανθρωπιστική βοήθεια για την αποκατάσταση και την ανοικοδόμηση σε μία πρώτη φάση. Λάβαμε υπόψη λοιπόν τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι 200 εκατομμύρια θα είναι διαθέσιμα πρόθεσμα μετά από, τις, από την κάλυψη και την αξιολόγηση των αναγκών θα υπάρξει μια διεθνής διάσκεψη για την IT. Νομίζω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα δώσαμε μια αρκετά σημαντική απάντηση. Ε, θα δοθεί βοήθεια και προς τη Δομινικανή Δημοκρατία Νομίζω ότι ένα πράγμα είναι να συλλέξουμε τα χρήματα, ένα δεύτερο πράγμα είναι να πάνε τα χρήματα σε αυτούς που πραγματικά τα χρειάζονται. Πρέπει να στοχεύσουμε σωστά τις ανάγκες της ανοικοδόμησης. Σύμφωνα με τα αιτήματα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη βοήθεια στη μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας και δυνάμεων αστυνομικών, θα ενισχύσουμε τη συνεισφορά μας και θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε προτάσεις για την παρέμβασή μας στον τομέα αυτό. Μετά από τη συνάντηση θα του Συμβουλίου χτες θα ακολουθήσει μια συνάντηση επιγόντως για θέματα τήρησης τάξης και θα δούμε αν υπάρχει δυνατότητα βοήθειας και μέσω της Ευρωπαϊκής Δύναμης Χωροφυλακής. Όλα αυτά θα αποφασιστούν τις επόμενες μέρες έτσι ώστε η αντίδρασή μας να είναι γρήγορη. Την επόμενη Δευτέρα θα συζητήσουμε το θέμα εκ νέου Πρόκειται για ένα θα έλεγα σημαντικό θέμα το οποίο θα δοκιμάσει τις δυνατότητες και τις επιδόσεις μας. Ο λαός της ΑΙΤΙΣ αλλά και οι ευρωπαϊκοί λαοί απαιτούν να υπάρξει μια γρήγορη και αποτελεσματική βοήθεια την οποία ελπίζουμε να χορηγήσουμε. Υπολογίζω στη βοήθειά σας, χαίρομαι που είμαι παρούσα σήμερα και σας μεταφέρω τις πληροφορίες αυτές και περιμένω τις πληροφορίες τις δικές σας. Ευχαριστώ κύριε Άστον. Το λόγο έχει εξ ονόμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο Επίτροπος Κάρελ Ντεχόχτ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου, ξεκινώντα να υπογραμμίσω την πρωτοφανή χρειά της καταστροφής και από πλευράς ανθρωπιστικού αντικτύπου, αλλά και από πλευράς επιπτώσεων στο σύνολο της χώρας. Γνωρίζετε ότι η ΑΕΤ είναι από τις πιο φτωχές χώρες του κόσμου σε μια χρόνια κατάσταση ευαισθησίας και εύθραυστη και οι ίδιες οι βασικές υποδομές και οι λειτουργίες της έχουν πολύ σοβαρά διαταραχθεί. Και η διεθνής κοινότητα επλήγει σκληρά, τα Ηνωμένα Έθνη και μη κυβερνητικέ ε, οργανώσεις και δικοί μας ε, υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακόμα αγνοούνται. Ε, πράγμα που εξηγεί τις δυσκολίες να οργανώσουμε την επιτόπου βοήθεια. Και το θέμα δεν είναι ε, ανικανότητα, αλλά έχει πληγεί και η διεθνή κοινότητα σημαντικά, γι' αυτό οι διαδικασίε ανακούφιση δεν ρέουν με τον τρόπο που κανεί θα επιθυμούσε. Ε, ωστόσο, ώρα με την ώρα αυτό βελτιώνεται. Με άλλα λόγια, λοιπόν, το θέμα δεν είναι μόνο να βοηθήσουμε να σωθούν ανθρώπινε ζωέ. Αυτό ε, θα πρέπει να σώσουμε μια χώρα ολόκληρη. Γι' αυτό και Είπα ότι εκπρόσωπος κάθε Άστον ε, συνεκάλεσε την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου. Πάρα πολύ χρήσιμο αυτό το εργαλείο για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Επιτρέψτε μου τώρα πάρα πολύ σύντομα να επιμείνω στις βασικές προκλήσεις. Πρώτον, ε, οι ανθρωπιστικέ ανάγκες τεράστιες που θα πρέπει να τι αντιμετωπίσουμε και γρήγορα κατεπίγουσα ιατρική φροντίδα, νερό, ε, υγιεινή, γιατί υπάρχουν κίνδυνοι ας πούμε ακόμα και για χολέρα. Ε, θα πρέπει να δοθεί στέγη και τροφή και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, χειρουργία, επεξεργασία υδάτων, στέγη, νερό, γενικά πρώτης ανάγκης βοήθεια. Οι προτεραιότητες μας λοιπόν είναι να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες, να έχουμε μια καλύτερη εικόνα λεπτομερή των αναγκών και να οργανώσουμε την επιμελητία και τις ε, μεταφορές της βοήθειας, όλα αυτά στα πλαίσια των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. <coughs> Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι ε, είναι πολύ δύσκολο σε τέτοιου είδους ε, συνθήκες να οργανώνουμε την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας. Ήθελα να ε, τονίσω ότι λίγες ώρες ε, μετά το σεισμό, το ανθρωπιστικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΚΟ και η ΜΙΚ συνεργάστηκαν και συνεργαζόμαστε και με μια οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών και είμαστε σε επαφή με τον Τζον Χόλμς που είναι επίσης ένας αξιωματούχος του ΟΗΕ. Θα πρέπει να αποκατασταθούν οι βασικές κρατικές υποδομές και λειτουργίες. Πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να ξαναρχίσει να λειτουργεί η χώρα, όχι από πλευράς ε, κτηρίων και μόνο που έχουν καταρρεύσει πολλά κτίρια, αλλά αγνοούνται και πολλοί κρατικοί λειτουργοί, υψηλοί αξιωματούχοι και έχουν διατραφεί οι βασικέ κρατικέ λειτουργίε. Το, έχει υπόψη του το Συμβούλιο αυτό και ε, πολύ σύντομα θα αποσταλεί ομάδα ειδικών εμπειρογνωμόνων τη Ένωση για να καταγράψει τι βασικέ πολιτικέ ανάγκε του κράτου, τη κρατική μηχανή για να δοθεί η τεχνική και ουσιαστική λειτουργία και σε διπλωματικό επίπεδο μπορεί να γίνει αυτό, αλλά αυτό ξεπερνάει τα όρια της διπλωματίας. Τις επόμενες μέρες αυτό θα το δούμε όλο να οξύνεται και ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αντιδράσουμε και μαζί με το Συμβούλιο να έχουμε ρόλο ηγετικό στην αποκατάσταση των κρατικών δομών και υποδομών και της λειτουργίας, ε, όχι μόνο τα κτίρια στη συνέχεια αποκατάσταση ενοικοδόμηση της χώρας πέρα από την άμεση επίγουσα βοήθεια σε επόμενες εβδομάδες ε, πολλά σωστικά συνεργεία και ε, πολλοί από τους ε, ανθρώπους που βοηθούν αυτή τη στιγμή θα έχουν φύγει και υπάρχει ο κλασικός κίνδυνος μιας δεύτερης καταστροφής όταν θα έχουν αποχωρήσει οι πρώτες βοήθειες. Θα πρέπει λοιπόν μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα να υπάρχει ένα σχέδιο των Ηνωμένων Εθνών αποκατάσταση της χώρας με σωστό επιμερισμό εργασίας μεταξύ των θεσμών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών για να υπάρχει μια καλή ε, συνεργασία για την απτυξιακή βοήθεια, τη βοήθεια αποκατάστασης για να υπάρχει μια ομαλή και ταχεία μετάβαση στην, μετά την πρώτη περίοδο εποχή και προσβλέπουμε και στη συνεργασία όλων των κρατών μελών, όλες τις δεσμεύσεις μας για συνεργασία και αποτελεσματικότητα της βοήθειας να γίνουν πράξη. Και εδώ πραγματικά θα δοκιμαστεί η ισχύ και ο στένος μας. Και τελευταίο στοιχείο το οικονομικό, όπως είπε ήδη η πρόσωπος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει να διαδραματίσει εκεί πρωταγωνιστικό ρόλο. Καταρχάς βεβαίως από πλευράς ανθρωπιστικής βοήθειας, 30 εκατομμύρια ευρώ εκ των οποίων τα 22 είναι ε, πραγματικά νέοι πόροι πέρα από τις ε, ανθρωπιστικές μας υποχρεώσεις και δεσμεύσεις προς την ΑΕΤ. Και δεν είναι μόνο η ανθρωπιστική βοήθεια, σας είπα, η δημιουργία των κρατικών θεσμών, η αποκατάσταση του κράτους και 100 εκατομμύρια ευρώ ε, περίπου 50 από παλιούς πόρους και 50 εκατομμύρια από νέους πόρους. Και τώρα ε, ε, γίνεται λόγος και για 200 εκατομμύρια, ενώ οι Αμερικανοί μιλούν για δισεκατομμύρια, 10 δις ε, εκατομμύρια δολάρια. Είναι ένα ποσό το οποίο δεν μπορεί να καλύψει ο, ο προϋπολογισμός μας, αλλά θα γίνει μια διάσκεψη δωρητών και ε, θα προχωρήσουμε σε περισσότερα κονδύλια. Λοιπόν, αυτό είναι το πακέτο ή δέσμη μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρα από τις ε, συνεισφορές των κρατών μελών που ήδη καταβάλλονται θα καταβληθούν στο μέλλον. Όπως είπε η, δέσμοι μετρων της ευρωπαικης ενωσης τη εκπρόσωπος, θα μεταβώ εγώ στην περιοχή και στην ΑΕΤ και στη Δημοκρατία. Αύριο το πρωί ταξιδεύω για να έχω επαφές με τις αρχές και να προσπαθήσουμε να ξαναστήσουμε τους θεσμούς του κράτους και με τον Πρόεδρο και με τι μεγαλύτερε μη κυβερνητικέ οργανώσει που δραστηριοποιούνται εκεί. Θα πω και στη Δομινικανή Δημοκρατία. Είναι σημαντικό να δούμε και ε, τη γειτονική χώρα και η κυβέρνηση. Και βλέπουμε ήδη ότι στα σύνορα ε, υπάρχει κίνδυνος να ε, δημιουργηθούν κάποιες εντάσεις. Οπότε θα εδώ για τους ηθήνοντες και της Δομινικανής Δημοκρατίας. Αυτά νομίζω κύριε Πρόεδρε έχω να πω προς το παρόν. Ε, στη συνέχεια θα απαντήσω και ε, τη Δευτέρα το απόγευμα επιστρέφοντας στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ακολουθούν οι ομιλητές εξ ονόματος των πολιτικών τους ομάδων. Πρώτος από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ο κύριος Γκέι Μίτσελ. 1,5 λεπτό παρακαλώ. Um, Πρόεδρε, φαντάζομαι το σώμα μας θα θυμάται ότι έχουμε αγνοούμενους από το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ και νομίζω ότι είναι η στιγμή να σκεφτούμε όλους τους αγνοούμενους στην ΑΕΤ αυτή τη στιγμή. Ο τρόπος Τεχούτ μας είπε ότι θα επισκεφτεί τη χώρα και θα αναφέρει τα συμπεράσματά του όταν επιστρέψει τη Δευτέρα το απόγευμα στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Αυτό είναι ιδιαίτερα επικοδομητικό, αλλά μιλάμε εδώ για μια καταστροφή χωρίς προηγούμενο Νομίζω δεν είναι υπερβολή να πει κανεί κάτι τέτοιο για μια τέτοια χώρα. Και πρέπει εδώ να σχολιάσω κιόλα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να φανεί και να προβάλλει περισσότερο την παρέμβασή τη. Η Λιβατό εκπρόσωπο και αντιπρόεδρο τη Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει πιο, με μεγαλύτερη προβολή τη δράση εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ο μεγαλύτερο δωρητή ανθρωπιστική βοήθεια η Ευρωπαϊκή Ένωση παγκοσμίω, με 60% τη παγκόσμια ανθρωπιστική βοήθεια και επίσης έχουμε σοβαρές δωρές και βλέπουμε όμως και τη συμμετοχή του ΟΗΕ και τα νοσοκομεία που βρίσκονται υπό την αγίδα του ΟΗΕ. Θα έπρεπε λοιπόν η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι πιο προβεβλημένη, να υπάρχουν ίσως ε, ομάδες ε, που να είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν κατεπίγουσες ανάγκες και να μεταβούν στην περιοχή εφόσον υπάρχει κρίση. Μιλάμε εδώ για μια χώρα που γνωρίζει μια μεγαλύτερη ακόμη κρίση λόγω της φτώχειας που επικρατεί εκεί. Μην ξεχνάμε την ΑΕΤ λοιπόν ούτω ή άλλω. Αυτή τη στιγμή πρέπει να θυμηθούμε ότι οι συνθήκε ήταν δυσμενεί ούτω ή άλλω. Ευχαριστώ. Μίτσελ. Ευχαριστώ κύριε Μίτσελ. Εξ ονόματο των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, το λόγο έχει τώρα για δύο λεπτά η κυρία η αλλω ευχαριστω ευχαριστω κυριε μιτσελ εξ ονοματο των σοσιαλιστων και Μακάβαν. Um, thank you, Mr. Um, our today... Ευχαριστώ. Όλοι σκεφτόμαστε το ότι υφίσταται αυτή τη στιγμή η ΑΕΤ και κυρίως ο λαός της ΑΕΤ και τους στέλνουμε τα συλληπιτήριά μας. Μια τραγωδία. Όπως είπε ο Μίτσελ, μια τραγωδία σε μια χώρα όπου το 75% του κόσμου ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Αυτό δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε άλλο πια. Το κοινό των χωρών μας ανταποκρίθηκε με εξαιρετικό τρόπο στην πρόκληση 13 εκατομμύρια λίρες στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσα σε δυο 3 μέρες κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Το κοινό μας στηρίζει λοιπόν να συλλέξουμε αυτές τις δωρές για την ΑΕΤ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Άστον γιατί μπόρεσε να συντονίσει μια πολιτική απάντηση γρήγορα. Την εποχή που είχε γίνει το τσουνάμι ε, είδαμε ότι ο σωστός συντονισμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός, όσο σημαντικός όσο και ε, τα χρήματα που συλλέγονται. Το θέμα δεν είναι ποια σημαία έχουν τα χρήματα αυτά, αλλά θα πρέπει να συνεργαστούμε με τα Ηνωμένα Έθνη. Μακροπρόθεσμα, χαίρομαι που θα υπάρξει μια διάσκεψη δωρητριών χωρών για την IT. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα της IT να δούμε τι θα γίνει με το χρέος της ΑΕΤ. Ελπίζω το θέμα του χρέους της ΑΕΤ, η οποία χρωστάει περίπου ένα δις δολάρια σε διεθνείς ε, πιστοτικά ιδρύματα, ιδιαίτερα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο έδωσε 150 εκατομμύρια ένα δάνειο. Μπορούμε αυτά τα χρήματα να είναι χρήσιμα. Το θέμα δεν είναι να χρεωθεί η χώρα αυτή και να γίνει ακόμα πιο φτωχή για τα επόμενα 100 χρόνια. Ελπίζω να τα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Το θέμα των συνόρων με τη Δομινικανή Δημοκρατία έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία επίσης. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και ελπίζω όλοι μαζί να συντονίσουμε την ανταπόκρισή μας. Ευχαριστώ κύριε Μακάβαν. Εξ ονόματος των φιλελευθέρων τώρα το λόγο έχει για 1,5 λεπτό ο κύριος Άιλουαρντ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχηθώ στη Βαρόνια στον υπάτη εκπρόσωπο, στις μεγάλες προκλήσεις που θα έχει να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της θητείας. Να Ότι και είπαν και τα Ηνωμένα Έθνη ότι είναι η μεγαλύτερη καταστροφή των τελευταίων δέκα Και από πλευρά θυμάτων και από πλευρά καταστροφών. Αρχίζει να φτάνει η ανακουφιστική βοήθεια, αλλά βλέπουμε ότι είναι τεράστια τα προβλήματα για να φτάσει βοήθεια σε εκείνους που την έχουν περισσότερη ανάγκη. Η ασφάλεια, προβλήματα γραφειοκρατίας, προβλήματα επιμελητίας έχουν καταγράψει ΜΚΟ και τα προβλήματα στη βοήθεια επιδεινώνουν ακόμα την κατάσταση και η αιτινή είναι μεταξύ ζωής και θανάτου. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, να ανακουφιστεί αυτή η κατάσταση, το χάος. Χρειάζεται συνεργασία και συντονισμός. ΜΚΟ, κυβερνητικοί σχηματισμοί, ε, τοπικές αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται για την επίγουσα παροχή βοήθειας εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο. Είναι σαφές ότι χρειάζεται αμέσως μαζική ε, διεθνής υποστήριξη. Ε, τεράστια η αλληλεγγύη και η οικονομική συνεισφορά και των πολιτών. Πάνω από 420 εκατομμύρια ευρώ ανθρωπιστική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ήδη ανακοινωθεί. Αυτό δείχνει και ηγετική στάση και αλληλεγγύη, αλλά θα χρειαστεί σημαντικό συντονισμός. Και ελπίζω, κύριε Άστον, και εσείς και Επίτροπος Ντεχόχ να συνεργαστείτε στενά. Ακούμε ότι θα μεταβείτε και στην περιοχή. Είναι το πιο φτωχό κράτος στο δυτικό ημισφαίριο και μεγάλη προτεραιότητα η αποκατάσταση της χώρας. Χαίρομαι ε, για την καλή αρχή που αποτελούν τα 200 εκατομμύρια που ανακοινώνεται, αλλά ε, όσο περνάει καιρό και θα αποσπαστεί η προσοχή μα από την ΑΕΤ, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει στο ύψο των ευθυνών τη και των δεσμεύσεων. Ευχαριστώ. Για τρία λεπτά εξ ονόματο των Πρασίνων, η κυρία Ζολή. Πρόεδρε, κυρία Είπατε, πρόσωπε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή η νέα ανθρωπιστική κρίση που γνωρίζει η IT ίσως ξεπερνάει στο εύρος της όλες τις προηγούμενες. Νομίζω λοιπόν ότι θα είναι δύσκολο να βρούμε τα σωστά λόγια για να εκφράσουμε τη συμπόνια μας για τα θύματα, τους επιζώντες, τις οικογένειες που έχασαν τα μέλη τους, να εξηγήσουμε ότι τον πόνο τους τον καταλαβαίνουμε και να προσπαθήσουμε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα βίαιος, βέβαια, αλλά δεν εξηγεί και την έκταση των ζημιών παρόλα αυτά. Αυτό σημαίνει ότι η χρόνια ένδια ε, στην οποία ζούσε η ΑΕΤ είναι ένα από του βασικού λόγου που υπάρχει αυτή η κρίση σήμερα. Η διεθνή κοινότητα ω τώρα φάνηκε ανίκανη να φέρει αλλαγέ στη χώρα αυτή. Και μάλιστα τι επέβαλε επιπλέον πολιτικέ που ξέρουμε ότι σήμερα δεν έχουν δώσει αποτελέσματα. Ε, η διεθνή, τα διεθνή θεσμικά όργανα, η Ευρώπη επιβάρυναν την αδυναμία του κοινωνικού ιστού, τη οικονομία και των θεσμικών οργάνων τη ΑΕΤ. Τη δεκαετία του 70 στην επιστηστική βοήθεια η ΑΕΤ μάλλον ω προ τι επιστηστικές τη ανάγκε, κάλυπτε το 80% των αναγκών τη. Σήμερα εισάγει περισσότερο από το μισό των αναγκών τη. Αυτό σημαίνει ότι η τοπική παραγωγή έχει πληγεί. Η IT ε μέχρι τη, στιγμή, μέχρι τη στιγμή του σεισμού ήταν μια χώρα χωρίς πόρους και στερημένη από του πόρου του οποίου έπρεπε να έχει πρόσβαση. Θα πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε όσο δυνατόν περισσότερο την ΑΕΤ για να μπορέσει να ανακάμψει άμεσα. Από αυτήν την άποψη λοιπόν μπορούμε να εκφράσουμε την ε, θλίψη μας για τη δυσκολία της ανθρωπιστικής βοήθειας να φτάσει στη χώρα και θα πρέπει στο μέλλον να προβλέψουμε μια καινοτόμα προσέγγιση στην βοήθεια που θα προσφέρουμε. Και κυρίως να δούμε πώς θα σχεδιαστεί η αναπτυξική βοήθεια μακροπρόθεσμα να δούμε τι θεωρούμε ότι είναι ορθές προτεραιότητες. Γιατί όλα τα συμπεράσματα από την επιτόπια εμπειρία μας δείχνουν ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε τα κατάλληλα αποτελέσματα. Πρέπει να δούμε εμείς την τακτική που ακολουθούμε και την προσέγγιση μας, καθώς και την κινητοποίηση των, ε, ε, την εκταμείευση των κονδυλίων που και πόσο άμεσα μπορούμε να τα αποδεσμεύουμε για σκοπούς ανθρωπιστικής βοήθειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει για την ανθρωπαστική βοήθεια που θα αποστείλει στην ΑΕΤ 130 εκατομμύρια άμεσα και 200 εκατομμύρια για τις μακροπρόθεσμες ανάγκες. Αν συγκρίνουμε τους αριθμούς αυτούς με άλλα αριθμητικά στοιχεία, 157 δις δολάρια που οι τράπεζες της City και της Wall Street ε, ετοιμάζονται να καταβάλουν προκειμένου να καλύψουν ε, του χιλιάδε εργαζομένου που εκπροσωπούν πεζέ του, αυτό μπορεί να δείξει ακριβώ τι είδου ανθρωπιστική βοήθεια προσπαθούμε και εμεί να προβάλλουμε σε διεθνέ επίπεδο. Η κατεπίγουσα ανθρωπιστική βοήθεια είναι λοιπόν αναγκαία, αλλά δεν αρκεί. Δεν μπορεί τίποτε να υποταστήσει την ανθρωπιστική βοήθεια μακροπρόθεσμα και αυτήν δεν πρέπει να τη βιώνουν οι χώρε που είναι δικαιούχοι σαν ε, μια μορφή υποταγής. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τι χώρε που γνωρίζουν τι μεγαλύτερε δυσχέρειε, αλλά ταυτόχρονα να τι σεβόμαστε, να τι επιτρέπουμε να αποφελούνται από του ίδιου πόρου του. Και θα πρέπει να διευκολύνουμε την ΑΕΤ στο μέλλον. Να τι αποδώσουμε όσα τι οφείλουμε. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπατή Εκπρόσωπε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να βοηθήσουμε τα θύματα του σεισμού στην ΑΕΤ να ανοικοδομήσουν τη χώρα του. Μια χώρα που ήταν κατεστραμμένη πριν ακόμη τη χτυπήσει φυσική αυτή καταστροφή. Ευχαριστώ κύριε Ζολή. Εξ ονόματος των ε, συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, για ένα λεπτό κύριο κύριος Ντέβα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η σκέψη μας και η καρδιά μας τρέφεται στο λαό της Θα ήθελα να συγχαρώ την Βαρόνι Άστον και τον Κάρολ Ντεγκούχτ για αυτά τα οποία έχουν ήδη συμβεί. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα δοθούν χρήματα. Ήμουν... Ασχολήθηκα μάλλον πάρα πολύ στενά με το τσουνάμι στην Ινδονησία και στην Κίνα, πήγα στο σεισμό στην Τουρκία, είδα τι έγινε με σεισμού στην Κίνα και κάθε φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο ε, έχουμε πολλά προβλήματα σε επίπεδο υποδομών. Νερό στέλνουμε, τροφές στέλνουμε, αλλά οι υποδομές καταστρέφονται και δυσκολεύουν την ε, μεταφορά της βοήθειας. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε λοιπόν στον τομέα της ε, της βοήθειας αυτής της μεταφοράς. Ένα αεροπλανοφόρο έχει ελικόπτερα, έχει μονάδα παραγωγής πόσιμου ύδατος, έχει ιατρείο. Μήπως θα πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας να παρέχουμε τέτοιου είδους σκάφη τα οποία θα βοηθούν ιδιαίτερα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε αποτελεσματικά για να σώζουμε ζωές αμέσως μετά την καταστροφή. Από την Ενωτική Αριστερά για δύο λεπτά ο κύριος Λεγιαρίκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Πάτη, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να επαναλάβω πόσο μας έχει συγκλονίσει ε, η μοίρα ε, του λαού της ΑΕΤΗΣ. Μια εβδομάδα τώρα τα παιδιά της ΑΕΤΗΣ επιβιώνουν σε μια πραγματική κόλαση παγκόσμια αλληλεγγύη που πραγματικά είναι μου στην καρδιά μας αλλά θα πρέπει να ενισχυθεί, να έχει καλύτερο συντονισμό και να είναι μόνο στην υπηρεσία του λαού που πεθαίνει από τη δίψα, από την πείνα, δεν έχει στέγη, στερείται των βασικών ε, υπηρεσιών υγείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να αποδευσμεύσει κάποια κονδύλια, αλλά δεν μπορούμε να παραμείνουμε εκεί η ε, βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αυξηθεί σημαντικά και το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα να συνεισφέρει και αυτό τα ευρωπαϊκά ελαιονάσματα διατροφής θα πρέπει να σταλούν κατεπηγόντω στο λαό τη ΑΕΤ. Α είμαστε ειλικρινεί μεταξύ μα. Η Ήπειρο μα έχει πραγματικό χρέο απέναντι στην ΑΕΤ. Ένα χρέος αποκατάστασης μετά από τόσα χρόνια κυριαρχία και λαιλασία. Θα πρέπει να εξάγουμε όλα τα διδάγματα από τη δαιμονία που είχαμε ασκήσει στη χώρα αυτή, μαργαριτάρη της Καρεβικής. Τα διεθνή ιδρύματα ε, την οδήγησαν σε ασφυξία με επονίδιστα δάνεια και ακόμα πιο επονίδιστου του τόκους. Θα πρέπει αμέσως να ζητήσουμε χωρίς όρους διαγραφή του χρέους. Η ομάδα μας επιθυμεί η διάσκεψη που ε, θα γίνει προσεχώς στο Μόντρεαλ να προετοιμάσει μια διεθνή διάσκεψη αποζημίωσης, αποκατάστασης και αηφόρου ανάπτυξης της ΑΕΤ σε συνεργασία με τον αιτινό λαό. Η αποκατάσταση αυτή θα πρέπει να είναι υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών έτσι ώστε ο λαός της ΑΕΤ να ε, ανακτήσει την οικονομική και πολιτική του κυριαρχία. Η ΑΕΤ δεν επιτρέπεται να είναι ε, ένα παιχνίδι κυδαιμονίας κυριαρχίας μεταξύ μεγάλων δυνάμεων. Εμείς καλωσορίζουμε βεβαίως την αλληλεγγύη των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά αρνούμαστε και προειδοποιούμε αυτό η πραγματική καταστροφή να είναι ε, πρόφαση για τους βορειοαμερικανούς ηγέτες ε, να ε, καταλάβουν την ίσο, να τη διαχειριστούν, να τη διοικήσουν και να εγκαταστήσουν στρατιωτικές βάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι το παράδειγμα και να έχει στο μυαλό της μόνο το λαό και τα παιδιά της αιτής. Σας ευχαριστώ. Κολέγα. Ευχαριστώ, συνάδελφοι, εξ ονόματος της ομάδας Ελευθερία και Δημοκρατία. Για ένα λεπτό, κύριος Προβέρα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω την αίσθηση αλληλεγγύης μου απέναντι σε όλους αυτούς που χτυπήθηκαν τόσο άσχημα από αυτή τη φυσική καταστροφή. Τέτοιου είδους ε, καταστάσεις ε, με τεράστιες καταστροφές στον τομέα των υποδομών και με χιλιάδες νεκρούς είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν αν δεν αποκατασταθεί η τάξη και η δημόσια ασφάλεια. Η αδίποτε παρέμβαση καθίσταται ιδιαίτερος δύσκολη αν δεν υπάρξει σωστός συντονισμός για τη διανομή των ε, μέσων τα οποία έχουν συλλεγεί. Θα πρέπει να κατανοήσουμε το τι χρησιμεύει, για ποιον χρησιμεύει και πότε θα είναι χρήσιμο. Αυτό έχει σημασία. Ένα άλλο θέμα που πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι πολύ συχνά η γενεοδορία των δωρητών, είτε ιδιωτών είτε του δημοσίου, ε, γίνεται αντικείμενο κατάχρησης και πάρα πολλές ε, μορφές βοήθειας δεν πηγαίνουν σε αυτούς οι οποίοι την έχουν ανάγκη. Απαιτείται έλεγχος λοιπόν για να αντιμετωπιστούν οι κλοπές και οι καταχρήσεις ιδιαίτερα σε χώρες εύθραυστες με υψηλότατα επίπεδα διαφθοράς. Η Ευρώπη ελπίζω να πετύχει προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ και ολοκληρώνεται ο γύρος των ομιλητών εξ ονόματος των ομάδων τους με τον κύριο Γκριφίν για 1,5 λεπτό εξ ονόματος το μη εγγεγραμμένων. Κύριε Πρόεδρε, είναι ο η που βλέπουμε από την ΑΕΤ. Το μόνο που μπορούμε να αισθανθούμε είναι συμπόνια για τα αθώα θύματα αυτής της φυσικής καταστροφής. Όλοι εδώ πλειωνόμαστε καλά και είμαστε πρόθυμοι να δωρήσουμε. Εγώ θα μπορούσα να δωρήσω το σημερινό μου επίδομα για την IT και το ίδιο θα έπρεπε να κάνουν και όλοι οι υπόλοιποι ευρωβουλευτέ. Και μάλιστα ε, και οι δικοί μα εκλογέ με του φόρου του μπορούν να στηρίξουν την ανθρωπιστική βοήθεια. Αλλά και οι βιομηχανίε μα, οι τράπεζέ μα θα πρέπει να στηρίξουν την προσπάθειά μας, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις πιέσεις που ασκεί στην Ευρωπαϊκή Βιομηχανία και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Κλάδο δεν επιτρέπει αυτή την κινητοποίηση. Είναι συγκλονιστικές εικόνες που βλέπουμε από την ΑΕΤ και Πρόοροι θάνατοι σημειώθηκαν φέτος λόγω των συνθήκων φτώχειας και του κρύου που ε, επικρατούσε. Αλλά και στην Ευρώπη γνωρίζουμε ανάλογα φαινόμενα. Αυτό λοιπόν νομίζουμε ότι την πολιτική μας ηγεσία θα πρέπει να την κάνει να αισθάνεται ντροπή. Και αυτό το σκάνδαλο νομίζω δεν θα έχει την απαραίτητη προβολή στην Ευρώπη, ε, όπω θα μείνουν ανώνυμοι και οι ηλικιωμένοι που έχασαν τη ζωή του. Οι ζωέ λοιπόν χάνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι φόροι συνεχώ συλλέγονται. Και ε, βλέπουμε τι καταστροφέ που συμβαίνουν σε άλλε περιοχέ, χωρί να ασχολούμαστε με τα δικά μα προβλήματα στην Ευρώπη. Αυτό είναι υποκρισία. Έχουμε τη χριστιανική μα κληρονομιά βεβαίω, αλλά ποτέ δεν ακολουθούμε τι επιταγέ τη αιώνια αλήθεια που οι περισσότεροι εδώ αγνοούν. Ε, στον ε, Τιμόθεο 1.8 βλέπουμε ότι όποιος αρνείται την πίστη του είναι χειρότερος και από έναν άπιστο. Ε, και τώρα ακολουθούν οι υπόλοιποι ομιλητές μεμονωμένοι. Η κυρία Στριφλέρ έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως ακούστηκε προηγουμένως η καταστροφή αυτή είχε πάρα πολύ μεγάλο μέγεθος λόγω της ισχυρότητας του σεισμού που θα οδηγήσει θα έλεγα σε ένα τεράστιο αριθμό νεκρών. Συγχαίρω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια γρήγορη και αποτελεσματική αντίδραση και για την υπόσχεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαθέσει μέχρι 429 εκατομμύρια ευρώ και για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών και μακροπρόθεσμα. Παρ' όλα αυτά οι Ευρωπαίοι αντιδρούν θα έλεγα αποσπασματικά και η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι ορατή, κάτι το οποίο έρχεται σε αντίθεση με την αποτελεσματικότητα της Αμερικανικής βοήθειας και αυτό μας κάνει να ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πρώτη δύναμη στον κόσμο που παρέχει βοήθεια σε τέτοιες καταστάσεις πρέπει εμείς να συντονίσουμε τις υπηρεσίες που έχουν τα διάφορα κράτη-μέλη, τα οποία χρησιμοποιούνται για να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Τα τελευταία γεγονότα δείχνουν ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η δυνατότητα αντίδρασης σε κρίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πολιτική άμυνα πρέπει να αναδιοργανωθεί, και προτείνω την πρόταση του Μισελ Μπαρνιέ από το 2006, έτοιμη που περιμένει να εφαρμοστεί, να υπάρξει μια ευρωπαϊκή δύναμη, Europaid, βοήθειας, και ο Βαν Ρομπί επίσης σήμερα είπε ότι πρέπει να υπάρξει μια τέτοια δύναμη άμεσης αντίδρασης. Μέσα σε λίγες μέρες οι Αμερικανοί ανέλαβαν ένα κυρίαρχο ρόλο στον τομέα αυτό. Είναι απαραίτητο να θυμίσουμε ότι ο ρόλος της κεντρικής και σφαιρικής Αντιμετώπιση ανήκει στις, στα Ηνωμένα Έθνη, τα οποία είναι σε καλύτερη θέση για να προχωρήσουν λοιπόν σε τέτοιου είδους ε, μορφές συντονισμού. Το θέμα δεν είναι βέβαια να ξοδευόμαστε σε τέτοιες ανόητες μάχες. Το θέμα είναι να υπάρχουν τα χρήματα και τα μέσα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πολίτες της έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν το τι ακριβώς συμβαίνει. Ευχαριστώ κύριο Στυρολιάν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. γιατί είναι καταραμένη, είναι καταδικασμένη στη δυστυχία ε, από την ανεξαρτησία και μετά, ε, εκτός από τις πολιτικές καταστροφές, έχει και τις θεομηνίες. Και ειδού σήμερα που αντιμετωπίζουμε μια ιστορική τραγωδία. Θάνατοι, τραυματίες, ανίποτη καταστροφή και ε, πλήρης κατάρρευση του κράτους. Θα πρέπει όμως να ξεπεράσουμε τη μυρολατρία και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, επιγόντως να βοηθήσει και ανθρωπιστικά και για την ενοικοδόμηση. Αυτό το οφείλουμε στους μεγάλους δεσμούς που έχουμε και ιστορικούς. Η παλιά ε, απικία και ε, αργότερα διπλωματική συνεργασία με τις ε, συμφωνίες Κοτονού που είναι προνομιούχος ε, γείτονα τη Ένωση τελικά γιατί έχουμε και τις ε, ε, άκρως απομακρυσμένες περιφέρειες που είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε την Ευρωπαϊκή Εξωτερική Υπηρεσία και τώρα κυρία Άστον είναι η πρώτη σας αποστολή αυτή. Όλες αυτός δείχνει ποιες είναι οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Πέρα από το κίνημα αλληλεγγύης της ε, οι Αμερικανοί μας θέτουν το ερώτημα κατά πόσο μπορούμε πράγματι να αντιδράσουμε. Ε, ευρωπαϊκός λοιπόν συντονισμό χρειάζεται με συνεισφορά των κρατών μελών ε, βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυστοκία στη συζήτηση αν θα στείλουμε ευρωπαϊκές δυνάμεις χωροφυλακής. είναι για το θέμα των Ηνωμένων Εθνών, αλλά τελικά ερχόμαστε να διαπιστώσουμε το εξή. Μήπω χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια αυτόνομη δομή που να έχει του απαραίτητου πόρου που χρειάζονται για την ανθρωπιστική βοήθεια για να μπορεί να παρεμβαίνει. Ε, Τέλο, η ανοικοδόμηση είναι τεράστια πρόκληση. Και πολλά τα εργοτάξια και πολιτικά και οικονομικά και περιβαλλοντικά και ε, μπορεί να είμαστε στο έτος μηδέν μιας νέας εποχής για την IT. Είναι ε, μεγάλο διακύβευμα και πρόκληση για την Ένωση που θα πρέπει να αποδειχθεί ηγετική δύναμη, αλλά να φαίνεται και τέτοια. Ευχαριστώ για 1,5 λεπτό. Ο κύριος Γκέρενς. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, οι ειδήσει των 8 μα το θυμίζουν κάθε βράδυ. Ο πόνο τη ΑΕΤ είναι αδύνατο να περιγραφεί με λόγια. Ίσως ο πόνος αυτό να μπορεί να συγκριθεί μόνο με τη συμπόνια που αισθάνεται σχεδόν όλο ο πλανήτη. Ε, η συμπόνια αυτή είναι σαφώ αυθόρμητη, αλλά δυστυχώ πρόσκαιρη παρόλο που είναι ειλικρινή. Σε 15 ημέρε, όταν τα μέσα μαζική ενημέρωση θα δώσουν προσοχή σε άλλα γεγονότα, θα σημάνει η στιγμή τη αλήθεια. Εάν δεν εξακολουθήσουμε τη δράση μα, οι Αιτινοί θα κινδυνεύσουν και πάλι να βρεθούν μόνοι, απομονωμένοι και εγκαταλειμμένοι στην τύχη του. Σε μια χώρα που τα πάντα πρέπει να γίνουν από την αρχή, ξεκινώντα από την αποκατάσταση και την ανοικοδόμηση, είναι σημαντικό ώστε οι φάσει αυτέ να οδηγήσουν σε μια πραγματική πολιτική ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ένα, εργαλείο, ένα κουτί εργαλείων ε, πλούσιων και μια σημαντική εμπειρία σε τέτοια θέματα. Γι' αυτό οι προκλήσει που αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία τη ΑΕΤ, που διθέτει καθόλου μέσα στη διαθεσή τη, πρέπει πραγματικά να, να, να αντιμετωπιστούν σαν να είναι η στιγμή τη αλήθεια και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει τι ερχόμενε ημέρε, μήνε και χρόνια να εργαστούμε κατά τρόπο αποτελεσματικό για να αντιμετωπίσουμε την, την αδιαφορία. Και αυτό μέσα σε μια προοπτική ανάκαμψη, προκειμένου να αποκατασταθούν οι συνθήκε ασφάλεια ασφάλεια και δημόσια τάξη και ώστε να υπάρχει συντονισμένη δράση σε μια χώρα όπου τα πάντα πλήγησαν από το σεισμό συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών ε, δομών. Μου φαίνεται λοιπόν συνετό να επιμένουμε σε μια σημαντική πτυχή. Η ανάκαμψη, η ανοικοδόμηση του Αιτινού κράτου θα πρέπει να είναι έργο των ίδιων των Αιτινών. Η δική του ανάπτυξη είναι το θέμα εδώ. Θα πρέπει λοιπόν να του βοηθήσουμε σε ένα πνεύμα εταιρική σχέση. Η Ευρώπη θα πρέπει στι διεθνεί διασκέψει να επιβεβαιώσει τη δράση που προβλέπει να αναπτύξει το θέμα αυτό και να πει ναι στην εταιρική σχέση και όχι στο τον πατερναλισμό και τον νέο αποκεκρατισμό. Ευχαριστώ κύριε Γκέρανς. Για ένα λεπτό ο κύριος Κόζουξνικ. Ναι, ε, Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Όλοι μας συμφωνούμε εδώ ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη τραγωδία των τελευταίων 200 ετών στην ΑΕΤ. Στη δική μας ομάδα των Ευρωπαίων συντηρητικών και μεταρρυθμιστών αλλά και στη χώρα μου, την Τσεχία, εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας τα θύματα. Παρ' όλα αυτά και παρόλη την έγκριση της συνθήκης της Λισαβόνας βλέπουμε ότι είμαστε ασυντόνιστοι και δεν έχουμε και ε, ουσιαστική δράση. Έχουμε πρόεδρο του Συμβουλίου, επίτροπο, ύπατη εκπρόσωπο και παρόλα αυτά ολιγορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορεί να αντιδράσει. Έχει αποκοιμηθεί. Τα κράτη-μέλη στέλνουν και οικονομική βοήθεια και υλικό. Εμείς τι κάνουμε. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό η κυρία Ήλτα Φιγκερέιντο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και εμείς συμφωνούμε με την έκφραση της θλίψης των υπολείπων συναδέλφων και βεβαίως εκφράζουμε τη συμπόνια μας για τον λαό της ΑΕΤ και την αλληλεγγύη μας προς αυτούς. Όμως δεν μπορούμε παρά να υπογραμμίσουμε ορισμένα στοιχεία τα οποία θεωρούμε καθοριστική σημασίας. Πρώτα απ' όλα απορρίπτουμε τη σκέψη ότι κάποιοι, κάποια ομάδα χωρών θα προσπαθήσουν να αποφεληθούν από αυτή την φυσική καταστροφή για να οδηγηθούν σε απεικιοκρατικές ενέργειες, όπως φαίνεται να γίνεται με την αποστολή ένοπλων στρατιωτών των ΗΠΑ ε, στη χώρα, ξεχνώντας τις συνθήκες φτώχειας τι οποίες ζει ο λαός της ΑΕΤ και που οδηγεί στην εκμετάλλευση των ανθρώπων αυτών από πολυεθνικές και από εξαγωγές ε, μαζικές άλλων χωρών προ αυτή τη χώρα, των ΗΠΑ ιδίω. Θα πρέπει λοιπόν η στήριξη ανθρωπιστική ανθρωπιστική μας βοήθεια να, γίνει, να δοθεί με προσοχή. Θα πρέπει να ανοικοδομηθεί η χώρα αυτή ώστε η τόλμη και το θάρρος των Αιτινών να αναγνωριστούν επιτέλους. Εδώ μιλάμε για Αφρικανούς οι οποίοι 800 τουλάχιστον χιλιάδες οδηγήθηκαν ως σκλάβοι στην ΑΕΤ και ήταν οι πρώτοι που έφεραν εις πέρα στην πρώτη κοινωνική επανάσταση στη Λατινική, στην Ήπειρο της Λατινικής Αμερικής με την ανεξαρτησία της χώρας. Θα πρέπει λοιπόν οι δράσεις μας να είναι άμεσες και συντονισμένες. Ευχαριστώ και τώρα 1,5 λεπτό η κυρία Αντζελίλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην Αττική διεξάγεται μια τραγωδία θα έλεγα φρικτή που προκλήθηκε από την φύση αλλά και από την απουσία των κρατικών υποδομών. Ένα κράτος που δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί ούτε κατελάχιστον την καταστροφή αυτή δεν μπορεί να διαχειριστεί τη βοήθεια προς τους πληθυσμούς οι οποίοι υφίστανται πολλά. Ο Ευθρός Σταυρός ήδη στις 25 ε, Ιανουαρίου ζητά να αντιδράσει με ενοποιημένο τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση για να τελειώσει το χάος και οι παρεμβάσεις οι οποίες δεν έχουν καμία χρησιμότητα. Θα πρέπει επίσης να συντονιστούν και τα κράτη-μέλη όπως το ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επίτροπη. Θα πρέπει να γίνει κυρίως μια προσπάθεια κυρία Άστον για τα παιδιά, ιδιαίτερα για τα ορφανά παιδιά που απαιτούν και ψυχολογική στήριξη γιατί αλλιώς θα καταδικαστούν στην φτώχεια και την εκμετάλλευση. Θα πρέπει η διεθνής κοινότητα να μην ε, οδηγηθεί ε, σε μια απλή θα έλεγα μορφή υιοθεσία των παιδιών της ΑΕΤΙΣ γιατί αυτό θα ήταν ουσιαστικά μια αναγκαστική εξορία ε, για τα παιδιά αυτά. Ο Ιταλός Υπουργών Εξωτερικών προτείνει την δημιουργία κάποιων δομών οικογενειακών στη συγκεκριμένη χώρα που θα βοηθήσει τα παιδιά αυτά να μεγαλώσουν με αξιοπρέπεια αλλά θα τους επιτρέπει να κάνουν και ταξίδια προς τον υπόλοιπο κόσμο σύντομα. Υπάρχει επίσης, και εδώ είναι η τελευταία μου ερώτηση, κάποιο σχέδιο για τη μείωση και κατάργηση του χρέους της χώρας αυτής. κυρία, Κρέτσο για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ. Όλος ο πλανήτης εκφράζει την αλληλεγγύη του και τη συμπόνια του για τα θύματα του καταστροφικού σεισμού στην Αίτη. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη άμεσης αντίδρασης στην κατάσταση αυτή. Θα πρέπει η βοήθειά μας να είναι στοχευμένη και αποτελεσματική. Βλέπουμε πώς οι διεθνείς ε, οργανώσεις έχουν ε, αντιδράσει τώρα, ιδίω οι φορείς του ΟΗΕ, αλλά κάποιε ε, μη κυβερνητικέ οργανώσει των κρατών μελών θα πρέπει, θα πρέπει επιχειρησιακέ δυνάμει τη Ευρωπαϊκή άμεσα να αναλάβουν δράση και Βλέπουμε σήμερα με το δράμα της ΑΕΤΗΣ ότι δεν αρκεί να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς να επιβιώσουν τώρα, αλλά θα πρέπει να στηρίξουμε και τις συνθήκες δημόσιας τάξης. Βρισκόμαστε σήμερα σε μια θέση όπου πολλοί άνθρωποι διαμαρτύρονται και κατηγορούν την ε, ε, επωνομαζόμενη κρυφή απεικιοκρατία την... λόγω της ανθρωπιστικής βοήθειας. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να στηρίξει την αξιοπιστία της στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην διαδικασία ανοικοδόμησης της ΑΕΤ. Θα πρέπει επίσης να στηρίξει τους κρατικούς φορείς της χώρας και θα πρέπει να φροντίσει για το καλό των κατοίκων, των λαών της ΑΕΤ και να δούμε κυρίω τι θα γίνει με τα ορφανά, τα ορφανά, τα παιδιά που έχασαν του γονεί του στη διάρκεια αυτή τη καταστροφή. Σου μινούτο την απαλάβρα. Ευχαριστώ. Ο κύριο Κόγουα, παρακαλώ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Ήπατη, πρόσωπο. Εδώ στο Κοινοβούλιο ακούμε διάφορες φωνές, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι η πολιτική αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε καλά συντονισμένη ήταν, ούτε επαρκής. Και τώρα θα πρέπει να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας προς τις ΜΚΟ και άλλους οργανισμούς που κάνουν τη δουλειά τους και γρήγορα και καλά. Εμείς θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Και έχω μία ερώτηση προς την υπάτη εκπρόσωπο, την κυρία Άστον. Είναι η πρώτη κατάσταση που έχετε να αντιμετωπίσετε, το πρώτο θέμα που έχετε να χειριστείτε. Πού καταλήγεται, ε, τι μπορούμε να βελτιώσουμε στο μέλλον, ποιο είναι το σημαντικότερο. Αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό. Ο συνάδελφος Φιλίπ Σουβά. Κυρία Άστον, φτάνει πια. Σε κάθε φυσική καταστροφή που συμβαίνει λέμε τα ίδια στέλνει το κάθε κράτο ξεχωριστά ένα αεροπλάνο ανθρωπιστική βοήθεια, οι Βέλγοι, οι Ιταλοί, οι Ισπανοί και ο καθένα από τη δική του τη γωνίτσα ε, βλέπει, βλέπουμε να, να οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα η κατάσταση αυτή. Δηλαδή επιτόπου να μην υπάρχει κανένα συντονισμό και απόλυτη αποδιοργάνωση. Πότε θα πάψουν όλα αυτά, πότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτέλου θα αναλάβει πραγματική δράση. Μόλι μα είπατε ότι όλα αυτά θα ήταν περίπλοκα. Αλλά μην το πείτε πάλι, γιατί υποτίθεται ότι τα πλάνα, τα σχέδια υπάρχουν. Ο κύριο Μπαρνιέ το 2006 είχε προτείνει τη δημιουργία μια ευρωπαϊκή δύναμη ε, προστασία των πολιτών βάσει τη οικειοθελού συμμετοχή των κρατών μελών. Και αυτό με την ομόφωνη άποψη των ε, κρατών μελών, προκειμένου να συνεργαστούν οι φορεί ανθρωπιστική βοήθεια των ε, κρατών μελών που ήδη υπάρχουν, να συντονίζονται, να εκπαιδεύονται μαζί, να υπάρχει ένα κοινό επιτελείο, κοινέ δυνάμει αντίδρασης. Είναι απλό κυρία Άστον. Και το θέμα είναι ότι πρέπει όλου να του πείσουμε όταν πιστούν ότι αυτό μόνο είναι λύση για το μέλλον. Τα είδαμε αυτά και μετά το τσουνάμι. Σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα εντωμεταξύ. Και ζυγίζω, σταθμίζω τα λόγια που σα λέω, διότι η αδράνεια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εγκληματική. Κυρία Άστον, διότι γιατί μάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχώ να επαναλαμβάνει τα ίδια σφάλματα. Κανείς βεβαίως δεν θέτει να αφιβόλω την ε, καλή σας πρόθεση, αλλά σήμερα εδώ πρέπει να δεσμευτείτε για τη δημιουργία αυτής της Ευρωπαϊκής Δύναμης Συντονισμού. Το Ευρωκοινοβούλιο θα σας ακολουθήσει και θα σας στηρίξει. Εάν έχετε ανάγκη από στήριξη, θα σας τη δώσουμε, θα σας βοηθήσουμε. Αλλά προς Θεού, προς Θεού πάψτε να μας μιλάτε για συντονισμό και επιτέλους φροντίστε να τον πραγματοποιήσετε αυτόν τον ε, συντονισμό πριν την επόμενη φυσική καταστροφή. Ευχαριστώ για μισή λεπτό. Το λόγο έχει ο κύριο Κάσμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν κάποιοι που ε, δρούν και κάποιοι που μιλούν για το τι θα κάνουν. Και συγχαίρω το Συμβούλιο και την Επιτροπή και την ύπατη εκπρόσωπο για τη δράση τους. Τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν προβλέψιμο. Μα ήταν τελείως αδιανόητο αυτό που συνέβη. Και ακούω εδώ φτηνά πολιτικά επιχειρήματα, μικροπολιτική κατά των κρατών μελών, κατά της υπά της εκπροσώπου και της Επιτροπής. Αυτή η έννοια του επειδή ε, πάνε και τους βοηθούν οι Αμερικανοί να τους βγάλουν από τα συντρίμια και να σώσουν τη ζωή, τι θα το κάνει στο χέρι, θα το κάνει στην άκρη. Όχι, δεν θέλω επικοιοκράτες. Μα υποφέρουν οι άνθρωποι και θα τους βοηθήσουμε επειδή θα διώξουμε αυτή τη χείρα βοηθείας. Ντροπή σας. Α συντονιστούμε, να, να αναλάβουν οι Αμερικανοί το συντονισμό αν πρόκειται να σώσει ζωέ. Τι ζωέ θέλουμε να σώσουμε. Ξεχάστε την πολιτική ρητόρια. Συγχαρητήρια, μπράβο για τα λεφτά που δεσμεύετε. Συγχαρητήρια, Βαρόνι Άστον, που δεν παίζετε αυτό το θέατρο να πηγαίνετε και να χρησιμοποιείτε ένα αέριο χώρο για να σας δούμε ότι είσαστε εκεί. Τι να το κάνουμε αυτό, δεν το χρειαζόμαστε καθόλου. Και γι' αυτό ε, έχω θυμώσει πραγματικά εξ ονόματο εκείνου που θέλουν τη βοήθεια να τους σώσουν. Ας συντονιστούμε με τους Αμερικανούς, με τον ΟΗΕ να βοηθήσουμε για να δοθεί η βοήθεια και σταματήσουμε τώρα να κάνουμε φτηνή μικροπολιτική. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Por un minuto tiene la palabra el Για 1,5 λεπτό η συνάδελφος Τούνον Χόενστάιν. Panie Przewodniczący, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να υποστηρίξω αυτά που μόλις είπε ο κύριος Ζουβά. Η ανθρωπιστική βοήθεια δεν είναι αρκετά συντονισμένη. Αλλά δεν θέλω να μιλήσω μόνο για την ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά και για την τεχνική υποστήριξη και την υποδομή και την αναπτυξιακή βοήθεια. Βεβαίως αυτές οι καταστροφές δεν είναι προβλέψιμες, αλλά γνωρίζαμε σε ποια δραματική κατάσταση βρισκόταν η ΑΕΤ έτσι και αλλιώς. Και δυστυχώς επλήγει και από αυτή τη τραγική θεομηνία. Γνωρίζαμε ποια είναι η πολιτική κατάσταση, οι κακές υποδομές στην IT. Και φυσικά θα μπορούσαν όλα αυτά να είναι καλύτερα αν είχαμε οργανώσει σωστά τη βοήθειά μας εκ των προτέρων και την ανθρωπιστική και τη γενικότερη και την αναπτυξιακή και τις υποδομές για να μπορούμε σήμερα να είμαστε σε καλύτερη μοίρα και να σώσουμε χιλιάδες ζωές. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Κυρία Άστον, στο Συμβούλιο που εργάζεστε προβλέπετε συγκεκριμένες δράσεις ακριβώς για να βεβαιωθείτε ότι θα υπάρχει συντονισμός μεμονωμένων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να είναι προς όφελος των τρίτων χωρών η βοήθεια αυτή. Θα ακολουθήσουμε την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει εμπειρία σε συγκεκριμένες χώρες και στη δική σας ε, με τρόπο πάρα πολύ αποτελεσματικό χορηγείτε τη βοήθεια και πολύ χρήσιμο θα ήταν ε, να ε, δοθούν αυτές οι πρακτικές και σε άλλες χώρες με λιγότερη παράδοση, με λιγότερη πείρα. Θα ήταν προς όφελος όρων για τις τρίτες χώρες η ανταλλαγή αυτών των πρακτικών και για την ανθρωπιστική βοήθεια και γενικότερα. Και θα είχαμε πιο συντονισμένη δράση. Ευχαριστώ κύριο Σασόλη για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Άστον. Μια τεράστια τραγωδία χτύπησε την ΑΕΤ τις τελευταίες μέρες και απαιτεί μια άμεση απάντηση. Έχουν ξεκινήσει αρκετές δραστηριότητες βοήθειας από πλευρά των μεμονωμένων κρατών μελών και υπάρχει θα έλεγα μια αρκετά υψηλή δόση ανταγωνισμού ανάμεσα στις διάφορες χώρες. Η Νέα Ευρώπη μέσω ημών θα πρέπει να προσπαθήσει να βοηθήσει άμεσα τον πληθυσμό γιατί ο σεισμός αυτός δυστυχώς χτύπησε την πιο φτωχή χώρα του δυτικού ημισφαιρίου, όπου το 80% του πληθυσμού ζει κάτω από το επίπεδο της ένδυας και ε, το 54% κάτω από το όριο της απόλυτης στόχιας όπως ορίζεται. Ιδιαίτερα οι ανήλικοι είναι οι πιο ευάλωτοι, οι πιο εύθραυστοι, ζουν χωρίς οικογένεια, χωρίς προστασία και χωρίς παρουσία κρατικών δομών. Και γι' αυτό θα ήθελα να προσκαλέσω την είπα το εκπρόσωπο να λάβει μέρος, να προσπαθήσει να καλύψει τις ανάγκες των, των παιδιών μέχρι την ηλικία των 10. Η Ευρώπη να προστατεύσει τα παιδιά αυτά. Πρέπει να προσπαθήσουμε να προσφέρουμε στα παιδιά αυτά για μια συγκεκριμένη περίοδο σύντομη περίοδο να τους προσφέρουμε φιλοξενία και να επιστρέψουν στην πατρίδα τους σε λίγο καιρό. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν, όλα αυτά είναι εύκολα και μπορούν να οργανωθούν από τα κράτη-μέλη. Έτσι θα απαντήσουμε στην απαραίτητη μορφή αλληλεγγύης η οποία πρέπει να υπάρξει και να αποφύγουμε επίσης και παράνομες δραστηριότητες εις βάρος των παιδιών. Μιλάμε για τα παιδιά, μιλάμε για ό,τι πιο πολύτιμο μπορούμε να προστατεύσουμε στην φτωχή αυτή χώρα. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό η κυρία Ανδρική Ένε, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τις τελευταίες ημέρες ακούσαμε πολλά παράπονα για την αναποτελεσματικότητα και την έλλειψη ταχείας απόκρισης ε, της κρίσης στην IT. Βλέπουμε η ανασφάλεια να αυξάνεται συνεχώς και ιδίω μεταξύ των, των επιβιωσάντων και να μην υπάρχουν τρόφιμα και νερό. Εδώ χρειάζεται να λύσουμε τα προβλήματα συντονισμού που έχουμε. Θα πρέπει να συντονιστούμε, να συνεργαστούμε και να επικρατήσουμε βεβαίω τη δράση διεθνών φορέων όπως κυβερνήσεων ή οργανώσεων πολιτών ή ε, ατόμων, μεμονωμένων παγκοσμίω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεταξύ εκείνων που εξέφρασαν την εγκάρδια αλληλεγγύη τους προ τον λαό της Αιτή. Και πάλι όμως πολλοί επέκριναν την ε, καθυστερημένη αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κρίση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως δεν είναι μόνο οι συναντήσεις και συνεδριάσεις της Βρυξέλλες. Οι κυβερνήσεις έχουν ήδη αποστείλει χιλιάδες ε, ευρώ για την βοήθεια στην ΑΕΤ και έχουν ήδη δεσμεύσει εκατομμύρια. Θα πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε στην μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βοήθεια στην ΑΕΤ, να ανοικοδομήσουμε τη χώρα, να τους ε, βοηθήσουμε τους ΑΕΤΙΝΟΥΣ να ξαναχτίσουν τη χώρα και τα σχολεία τους. Θα πρέπει να τους προσφέρουμε μια ομπρέλα προστασίας. Θα πρέπει η μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βοήθειά μας να μοιραστεί και να αποτελεσματικά και να γίνει αυτό με συντονισμό. Θα πρέπει η Επιτροπή και τα μέλη να συνεργαστούν ώστε το μισό ευρώ που μπορεί να συγκεντρωθεί να φροντίσουν να αποδεσμευτεί σωστά προ την σημαντική αυτή και ορθή κατεύθυνση και όλοι θα τη στηρίξουμε. Ευχαριστώ για 1,5 λεπτό, κύριο Γκερέρο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχά θα ήθελα να απευθύνω τα συλληπιτήρια και την αλληλεγγύη μου προς το λαό της ΑΕΤΗΣ που τόσο σφοδρά επλήγει από τη θεομηνία αυτή. Εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είμαστε στρατιωτική δύναμη, ούτε θέλουμε να είμαστε στρατιωτική υπερδύναμη. Είμαστε μια παγκόσμια δύναμη από το κοινωνικό μας μοντέλο. Και δύναμη είμαστε και θέλουμε να παραμείνουμε με την αναπτυξιακή μας συνεργασία και με τη βοήθεια που παρέχουμε την ανθρωπιστική. Σήμερα η θεομηνία και η καταστροφή στην ΑΕΤ αποτελεί πρόκληση για τους νέους θεσμούς που προέκυψαν από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Σήμερα είναι η ώρα της ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά πολύ σύντομα θα έρθει η ώρα της ανοικοδόμησης, της ε, βοήθειας στην ανάπτυξη και στη ε, δημιουργία θεσμών και κυβέρνησης. Και θα πρέπει να απαντήσουμε με μία φωνή σε αυτά που περιμένει από εμάς ε, ο λαός της ΑΕΤ θα πρέπει, είπατε, εκπρόσωπος να συνεργαστεί αρμονικά με τον ε, ε, Επίτροπο για την Ανάπτυξη και την Ανθρωπιστική Βοήθεια. Γιατί χρειάζεται κοινή δράση για να υπάρχει καλύτερο συντονισμό των ε, κρατικών βοηθειών, για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, για να έχουμε μία φωνή ευρωπαϊκή που να ακούγεται στον κόσμο και να είναι διακριτή και να αναποκρινόμαστε σε αυτά που περιμένει από εμά ο κόσμο. Υποστήριξη στην ανθρωπιστική κρίση, όθηση για την ανάπτυξη. Σήμερα στην Αιτία, αύριο δεν ξέρω πού και μεθαύριο παντού, απανταχού τη γη. Ευχαριστώ. Ρίκε. Για 1,5 λεπτό τώρα ο κύριος Jim Higgins. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μία από τις φτωχότερες χώρες στον κόσμο μέσα σε 15 δευτερόλεπτα καταστράφηκε. Είναι θύμα των φυσικών καταστροφών, είναι θύμα της δικτατορίας, είναι θύμα της διαφθοράς και εκατοντάδες χιλιάδες αυτή τη στιγμή είναι αγνοούμενοι οι Ηνωμένε Πολιτείε προσπαθούν, τα Ηνωμένα Έθνη λίγο λιγότερο από ό,τι φαίνεται, αλλά θα συμφωνήσω με τον κύριο Κάσμαν ότι η απάντησή μας δεν ήταν η καλύτερη και απλά παρακολουθούμε αυτά που έκαναν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Τα επιμελητιακά προβλήματα θα ξεπεραστούν το πόσιμο νερό, η κυκλοφορία, οι μεταφορές λοιπά θα βελτιωθούν. Αυτό που απαιτείται όμως είναι μια πλήρως λειτουργούσα δημοκρατία με την οικονομία να την συνοδεύει και να τη φροντίζει θα χρειαστούν προσπάθειες για πολλά χρόνια και όχι μόνο τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες. Το νέο θα φύγει από τις οθόνες της τηλεόρασης, θα παραμείνει ένα για λίγες μέρες, θα γίνει τρία σε λίγες εβδομάδες και στο τέλος θα χαθεί. Θυμίζω ότι το 2008 ε, καταστράφηκε πάλι η IT μετά από δύο πάρα πολύ ισχυρούς τυφώνες Είχαμε υποσχεθεί 600 εκατομμύρια ε, ε, ευρώ και δόθηκαν ελάχιστα τελικά στο τέλος. Και τίποτα δεν είχε σαν στόχο την ανάπτυξη της χώρας αυτής, τη σωστή ανάπτυξή της. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια σαφή στρατηγική έτσι ώστε η ΑΕΤ να γίνει μια περήφανη, ανεξάρτητη και δημοκρατική οντότητα που δεν είναι σήμερα και αυτό έχει συμβάλει στη σημερινή καταστροφή. Ευχαριστώ κύριε Χέγγιν Σογκουαλτιέρη για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. ανθρωπιστική καταστροφή χωρίς προηγούμενο στην ΑΕΤ μας συγκινεί βαθύτατα και επιβάλλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεισφέρει όσο μπορεί καλύτερα με όλα τα μέσα που διαθέτει. Σε οικονομικό επίπεδο έγιναν σημαντικά βήματα προόδου τις τελευταίες ημέρες. Αυτό το οποίο μένει ακόμα είναι οι άλλες πλευρές της ευρωπαϊκής απάντησης στην κρίση το θέμα δεν είναι η εικόνα και εγώ συμφωνώ, αλλά να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στην ουσία, όπως είπε η κυρία Άστον. Ο κεντρικός ρόλος της Μινουστά, της αδυνάμεως των Ηνωμένων Εθνών και σε επίπεδο πολιτικής προστασίας και σε επίπεδο ασφάλειας θα έλεγα μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμος και δεν χρειάζεται αυτόνομη παρέμβαση από πλευράς μας. Ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών είναι κεντρικός και πρέπει να το θυμίσω αυτό προς τον κύριο Ζούβα. Υπάρχουν υπηρεσίες σε διεθνές επίπεδο που ασχολούνται με τα θέματα της ασφαλείας, με τα θέματα της τήρησης της τάξης και της επιμελητίας γενικότερα. Αυτό το οποίο θα είναι χρήσιμο να καταλάβουμε μετά από αυτά που ακούσαμε και από αυτά που θα ακούσουμε από την είπα του εκπρόσωπο είναι πώς ανταποκρίνονται το MIC και το Situation Center της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συντονίζουν τη βοήθεια την κοινωνική. Τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους είναι ικανά, είναι αρκετά, είναι κατάλληλα τα μέσα αυτά. Θα μπορέσουν να βοηθήσουν, θα μπορέσουν να βοηθήσουν και τους συμπολίτε μας σε προξενικό επίπεδο που ατυχώς βρίσκονται εκεί Στιάει Ο κύριος Σβέρ για ένα λεπτό. Είπα το όνομα σας σωστά. Κύριος Σβέρ. Σβέρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμα Μέλη, κυρία Άστον, θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου ε, προς το λαό της ΑΕΤΗΣ. Ταυτόχρονα θα ήθελα να συγχαρώ όμως και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα γιατί αντέδρασαν σχετικά θετικά. Ανησυχώ βέβαια και εγώ όπως και άλλοι βουλευτές για το έγκαιρο της ε, παρέμβασής μας. Έχει σημασία να είμαστε παρόντες εκεί ε, στον τόπο της τραγωδίας για πολλούς λόγους. Ορισμένοι λέγουν ότι μπορεί να θεωρηθεί νεοαπικιοκρατία η παρουσία στρατού εκεί. Μα αυτό είναι άδικο. Στη διεθνή διάσκεψη για την ΑΕΤ θα πρέπει να ορίσουμε τα μακροπρόθεσμα μέτρα για να ξαναστήσουμε τους ε, κρατικούς θεσμούς, να μπορούν να λειτουργούν μόνοι τους, να βοηθήσουμε για τα σχολεία, για την υγεία, ε, όλη την κρατική υποδομή, έτσι ώστε η ΑΕΤ να γίνει πιο σταθερή χώρα. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα είμαι αρκετά αυστηρό με το του ΙΑΗ γενικώ και με το χρόνο. Παρακαλώ, όταν λέμε ένα λεπτό, ένα λεπτό. Η κυρία Μουνής για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της ηγετικής θέσης και του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι για την άμεση κατεπίγουσα ανθρωπιστική βοήθεια αλλά και πιο μακροπρόθεσμα για την ανοικοδόμηση σε συνεργασία με την κυβέρνηση της ΑΕΤ που είναι αρκετά εύθραυστη χώρα για να την ε, κλονίσουμε ακόμα περισσότερο ε, διαχειριζόμενοι διεθνείς οργανισμοί τη χώρα και υποκαθιστώντας τις τοπικές αρχές και τις κρατικές αρχές. Αναγνωρίζω ότι η Ισπανική Προεδρία αντέδρασε γρήγορα και στο συντονισμό και στη ε, διάθεση των μέσων που είχε η Ισπανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι ο πρώτος Ευρωπαίος δωρητής στην περιοχή, όχι μόνο στη Λατινική Αμερική και στην Αϊτή την ίδια. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Σαρνές για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κυρία Άστον, η πολιτική είναι κυρίω συμβολικά πρόσωπα. Γι' αυτό δεν νομίζω ότι πρέπει να είστε εδώ, αλλά στην ΑΕΤ. Και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να πάτε στι ΗΠΑ, αλλά απευθεία στην ΑΕΤ. Έχω επίση την εντύπωση, και το λέω αυτό με μεγάλη θλίψη, έχω την αίσθηση ότι δεν έχετε καταλάβει τι διαστάσει του συμβάντο, της αποτρόπη αυτή τη τραγωδία. Ποτέ η Ευρώπη δεν φάνηκε τόσο απούσα σε μια τόσο μεγάλη καταστροφή. Είμαστε πρώτοι δωρητέ, αλλά δεν υπάρχουμε, δεν φαινόμαστε. Και μια δεύτερη αίσθηση. Όσο περισσότερο έχουμε διορισμού, όσο περισσότερο δημιουργούμε θέσει και τίτλου, όλο και λιγότερο φαίνεται να είμαστε υπαρκτοί και αυτό θα πρέπει να μα απασχολήσει. Πόσε καταστροφέ θα πρέπει ακόμη να ζήσουμε, προκειμένου οι υπεύθυνοι τη Ευρωπαϊκή Ένωση επιτέλου να φανούν στο ύψο των ευθυνών του, των καθηκόντων του. Στο τραπέζι έχουμε ε, μια έκθεση του Μισελ Μπαρνιά το 2006. Τι περιμένουμε για να την εγκρίνουμε, τι περιμένετε για να την εφαρμόσετε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νίκολσον για ένα λεπτό. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα πρέπει να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας προς εκείνους που έχασαν τις ζωές τους και το λαό της ΑΕΤΗΣ ε, και ε, τους εργαζομένους των Εθνών και τους επιζήσαντες. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια προσπάθεια καλή και καλά συντονισμένη. Τίποτα, μα τίποτα δεν θα πρέπει να σταθεί εμπόδιο σε αυτό. Εγώ καλωσορίζω τη δέσμευση που κάναμε στην Ευρώπη για ε, να βοηθήσουμε και ελπίζω να δοθεί συνέχεια. Με συγκίνησε αυτό που ακούστηκε. Τι θα γίνει σε δύο εβδομάδες όταν θα σταματήσει ο τύπος να ενδιαφέρεται και οι ειδήσει. Ο κόσμος τι θα κάνει. Γι' αυτό θα πρέπει να ξαναχτιστεί η IT και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Τώρα το πιο σημαντικό είναι να δοθεί η βοήθεια στο λαό που υποφέρει επιτόπου. Και πρέπει να σας πω κύριε Πρόεδρε ότι θα συμφωνήσω απολύτως με αυτά που είπε προηγουμένως ο κύριος Κάσμαν. Είναι πολύ σημαντικό για να πέφτουμε σε μικροπολιτική. Ο κύριος ε, Γιάννης για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα μερικά δευτερόλεπτα μόνο να σας πω θέλω να συγχαρώ την υπάτη εκπρόσωπο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την εναρσόμενη Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ταχύτητα, την ε, ακρίβεια, το συντονισμό και τις προσπάθειες ε, που κατέβαλα. Βέβαια δεν είχαν την ε, κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης που είχαν 10.000 Αμερικανοί πεζοναύτες, αλλά πολύ γρήγορα αντέδρασαν και πολύ αποτελεσματικά. Σας δώσω ένα στοιχείο μόνο που δεν ακούστηκε ακόμα. στις 78 ώρες το 50% των ανθρώπων που σώθηκαν ήταν από Ευρωπαίους. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρίση, ένα λεπτό. Το είπε ήδη η κυρία Ζολή. Υπάρχουν καταστάσεις και συνθήκες όπου οι αριθμοί δεν έχουν πια νόημα, είναι περίτη. Δύο εκατομμύρια πρόσφυγες, πάνω των 100.000 νεκροί, μια πρωτεύουσα που έχει καταστραφεί, έχει σβήσει από το χάρτη πια. Το θέμα είναι πώς θα θάψουμε τους νεκρούς, θα θρέψουμε τους ε, εν ζωή και θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε. Κάθε χώρα ξεκίνησε το ταχύτερο δυνατόν με τα μέσα που έχει, με τους ανθρώπους που έχει. Η προσπάθεια που έχει γίνει μέχρι τώρα είναι εθνική βοήθεια. Η Ευρώπη τώρα θα πρέπει να πάρει τη σκητάλη και να προχωρήσει σε αυτό το οποίο ζητάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και αρκετό καιρό, δηλαδή τη δημιουργία ενός σώματος ε, Ευρωπαίων που θα βοηθήσουν στον τομέα της πολιτικής άμυνας, EU Force που ξεκίνησε με τον Γκί ε, στα παλιότερα, η ιδέα του Μπαρνιέ το 2006, Όλα αυτά θα βοηθήσουν να δράσουμε από κοινού και με μεγάλη ταχύτητα. Έχω την εντύπωση ότι αυτό που απαιτείται είναι η διαφάνεια και η σωστή στόχευση της βοήθειας απαιτείται να υπάρξουν αυτές οι δύο προϋποθέσεις. Η κατάσταση βέβαια είναι τρομερή. Βλέπουμε τα ερήπια και θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα από ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της ΚΕΠΑ δημιουργήθηκε και για να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους καταστάσεις και προβλέπεται να υπάρχουν ε, δομές που θα αντιμετωπίζουν τέτοιες κρίσεις και τέτοιες τεράστιες φυσικές καταστροφές. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε σε τέτοιου είδους καταστροφές. Άλλωστε και στην Ευρώπη πολλές φορές συμβαίνουν σημαντικές φυσικές καταστροφές. Δυστυχώς όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ανταποκρίνεται. Ευτυχώς στην Ευρώπη δεν έχουμε τέτοιες φυσικές καταστροφές ενώ τέτοιου μεγέθους. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα μας για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που υποφέρουν σήμερα. Ο κύριος Μπαλκίτης είναι εδώ. κύριε Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Άστον, κύριε Επίτροπε, μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνα, δυστυχώς τώρα αντιμετωπίζουμε μια καταστροφή που ουδέποτε έχουμε γνωρίσει τέτοια κλίμακα. Θα πρέπει λοιπόν το πρόσωπο που κατέχει το αξίωμα του είπατε εκπροσώπου να αναλάβει τα καθήκοντά του αμέσως. Βεβαίως εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάποιες δυσκολίες. Σαφώς στο μέλλον θα χρειαστούμε καλύτερα εξοπλισμένη και εκπαιδευμένη δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενδεχομένως σε συνδυασμό με τον ΟΗΕ που να λαμβάνει μέρος σε τέτοιες διαδικασίες διάσωσης αλλά Ταυτόχρονα η βοήθεια που έχουμε υποσχεθεί είναι το σημαντικότερο πώς θα εκταμιευθεί ακριβώς και πώς θα μοιραστεί. Θα πρέπει λοιπόν να προβλέψουμε κονδύλια για, τα, για το έργο ανοικοδόμησης της IT. Έχετε το λόγο. Uh, Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Ανυπομονούσα να φτάσω στο Κοινοβούλιο για να ακούσω τις απόψεις σας και καταλαβαίνω και την ε, ανησυχία και την απογοήτευση που κάποιοι συνάδελφοι στάνονται διότι θα μπορούσαν πολλά να έχουν γίνει καλύτερα. Πολλοί βουλευτέ ρωτούν τι γίνεται με την προβολή και το συντονισμό μας. Δεν υπάρχει θέμα ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται πιο κοντά στη χώρα και έχουν και τις δυνατότητες να κινητοποιηθούν άμεσα. Βεβαίω, η εικόνα που θα βλέπετε στι τηλεοπτικέ οθόνε θα είναι κυρίω αυτή των Αμερικανών. Όμω συνεργαζόμαστε στενά με τι ΗΠΑ και αυτό είναι ένα σημαντικό μέρο τη δράση μα και τη σημερινή και τη μελλοντική. Και ένα άλλο ερώτημα είναι ότι ήδη το βράδυ του σεισμού είχαμε αποφασίσει να κινητοποιήσουμε δυνάμει όσο τα δυνατόν συντομότερα. 21 κράτη-μέλη κινητοποιήθηκαν αμέσω για να ανταποκριθούν στι ανάγκε. Και εργαστήκαμε και στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. Συναντήθηκαν εκπρόσωποι αμέσω για πρώτη φορά Και στις 8 αυτό, αυτές οι μέρες πριν την ακροασή μου ε, ε, στείλαμε 80 ανθρώπους, 5 ομάδες διάσωσης, ε, μέλη προσωπικού, 14 ιατρικές ομάδες και ομάδες καθαρισμού, 6 τουλάχιστον. προσπαθήσαμε να κινηθούμε στο δυνατόν ταχύτερα και τα κράτη-μέλη αποδίδουν φόρο τιμή στο δικό μα έργο και εμεί εκφράζουμε την ικανοποίησή μα στα στελέχη που ε, εργάζονται νυχθημερών πολλέ φορέ για να συντονίσουν όλε αυτέ τι προσπάθειε. Ε, αγαπητοί βουλευτέ, ε, το θέμα είναι ότι ο ΙΕ έχει παρουσία επιτόπου και ο Γενικό Γραμματέα Κίμων έχει αναγνωρίσει την επιτυχία των προσπαθειών μα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αν εγώ επισκεφτώ την ΑΕΤ, το μόνο που θα κατανοώ είναι να καταλάβω πολύτιμο χώρο. Όταν αναζητείται χώρο προσγείωση για τα αεροπλάνα που δεν μπορούν για την ώρα να προσγειωθούν, διότι είναι ασφαλές, δεν είναι αρκετά ασφαλέ το αεροδρόμιο. Δεν είμαι πυροσβέστης, δεν είμαι μαχητής και δικός μου ρόλος είναι να συντονίσω τις προσπάθειες και να προσπαθήσουμε η ομάδα για την ε, άμυνα της ΑΕΤ να συντονιστεί με αυτή των ΗΠΑ ώστε να καταβάλουμε το μέγιστα για να βελτιώσουμε την κατάσταση επιτόπου. Και με κυβερνητικές οργανώσεις και οι εργαζόμενοι ήδη στην ΑΕΤ γνωρίζουν ότι η καταστροφή είναι τεράστια και ΙΕ ήδη έχει χάσει πολλά μέλη του προσωπικού του. Έχει μειωθεί λοιπόν η δυνατότητα απόκριση, το ίδιο και τι μη κυβερνητικέ οργανώσει. Γιατί έχουν πεθάνει ακριβώ άνθρωποι. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν και το έχετε δει και εσεί στι οθόνε σα όπω και εμεί. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι απελπισμένοι και ζητούν βοήθεια και αναρωτιούνται πού βρίσκεται αυτή η βοήθεια. Το να φτάσει η βοήθεια λοιπόν σε αυτέ τι συνθήκε ήταν ιδιαίτερα δυσχερέ και Πολλοί είναι οι άνθρωποι που εργάστηκαν ε, ασταμάτητα και αδιαλείπτω για να το καταφέρουν αυτό. Ξεκινάει η βοήθεια, πηγαίνει στην ΑΕΤ, αλλά μην έχετε για κανένα μια στιγμή αμφιβολία ότι τα πράγματα επιτόπου είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εάν πήγαν καλά τα πράγματα, ναι. Εάν είμαι ικανοποιημένη, όχι. Όταν ξεκίνησα την πρώτη εβδομάδα ανάληψη των καθηκόντων μου, σα το λέω ξεκάθαρα. Σα ακούω και ακούω και την απογοήτευσή σα και την ε, συμμερίζομαι και έχετε δίκιο να με επικρίνετε ότι τα πράγματα δεν ήταν τόσο καλά όσο θα μπορούσαν να γίνουν στο μέλλον. Έχετε δίκιο. Μπορούν και οφείλουν να γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Αλλά αυτό που κάνω είναι να παρακολουθώ τι γίνεται και να μάθω από τώρα τα διδάγματα για το μέλλον. ώστε στο μέλλον να ξέρουμε τι να κάνουμε. Τίποτε δεν θα το παραβλέψουμε. Αλλά δεν θα μειώσω και το, τη σημασία του έργου που έχει γίνει ω τώρα, που είναι σοβαρό και τεράστιο. Και σήμερα και ώρα με την ώρα. Ε, Πάντω οι βουλευτέ έχουν έχουν δίκιο όταν λένε ότι πρέπει να είμαστε εκεί και σωματικά και ε, ως προς την ε, βοήθεια που θα δώσουμε. Σαφώς θα πρέπει να έχουμε και τεχνικό προσωπικό και σαφώς θα πρέπει να φροντίσουμε οι αιτινοί ε, να έχουν μαζί μας μια εταιρική σχέση ώστε να μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Χρειάζεται υποδομές η χώρα, χρειάζεται ανοικοδόμηση. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ο ρόλος του ΟΗΕ αναγνωρίζεται και ότι μπορεί να φέρει πέρα στο έργο του το προσωπικό του ΟΗΕ όπως πρέπει. Οι Ηνωμένε Πολιτείε και ο Υπουργό Κλίντον και ο ΙΕ θα συνομιλήσουν, θα συνομιλήσουν τα μέλη του ΟΗΕ, ο Γενικό Γραμματέα, με του εκπροσώπου τη Αμερικανική κυβέρνηση για να καθορίσουν ένα δρόμο για το μέλλον. Αυτό θα είναι τεράστια σημασία. Και βεβαίω να πούμε πώ έχουν τα πράγματα και στην πράξη. Όπω είπαν πολλοί βουλευτέ, εδώ μιλάμε για μια χώρα που το 70% των ανθρώπων ήδη ζούσαν κάτω από το κατόφλι τη φτώχεια. Και είναι σημαντικό, όπω κάποιο είπε, τα παιδιά, τα ορφανά μετά από την πρόσφατη καταστροφή να τέχουν τις απαραίτητες περίθαλψη. Επίση να δούμε τι θα γίνει με την μακροπρόθεσμη στήριξη. Λίγα λόγια τελευταία λόγια για τις υποδομές αυτή τη στιγμή. Τα νοσοκομεία, ο ηλεκτρισμός, οι επικοινωνίες, το νερό, τα αεροδρόμια και οι υποδομές γενικώ έχουν καταστραφεί. Τα βασικά κτίρια, το Προεδρικό Μέγαρο, το Κοινοβούλιο, τα Υπουργεία των Οικονομικών, της Δικαιοσύνης, του κυβερνητικού σχεδιασμού και των εσωτερικών έχουν πληγεί σοβαρά. Πολλά τελέχη τη κυβέρνηση αγνοούνται και δεν λειτουργούν οι κυβερνητικέ δομέ. Όπω υπόθηκε, μιλάμε για μια από τι φτωχότερε χώρε ήδη στον κόσμο. Και ακριβώ επειδή πρέπει να ε, δημιουργήσουμε ξανά αυτέ τι υποδομέ, σα βεβαιώνω ότι θα δείξουμε όλη την απαραίτητη δέσμευση για να το πετύχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Και τέλος ο κύριος ε, Ντεγκούτ. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να πω στον κύριο Λεγιαρίκα που μας λέει να στείλουμε τα πλεονάσματα τροφίμων της Ένωσης ότι δεν είναι η προσέγγιση αυτή η δική μας για το λόγο ότι προτιμά η Ευρωπαϊκή Ένωση να αγοράσει τα προϊόντα στην περιοχή αυτό φροντίζουμε να κοιτάμε παρά να στέλνουμε τα δικά μας πλεονάσματα στην ΑΕΤ. Το δεύτερο, ε, το όλο ζήτημα του συντονισμού και της πολιτικής προστασίας κτλ. Θα ήθελα να σας πω τα εξής τρία. Πρώτον, η πολιτική προστασία είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Και όλες οι πρωτοβουλίες για συντονισμό θα πρέπει να βασίζονται σε αυτό το ε, γεγονός. Αυτό το προτείνει βέβαια και η έκθεση Μπαρνιέ. Γνωρίζουμε ποια είναι η πρόταση της έκθεση Μπαρνιέ, αλλά παραμένει αρμοδιότητα των κρατών μελών και όχι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά πάντα την πολιτική προστασία και το συντονισμό, από το τσουνάμι του 2004, η πολιτική προστασία συντονίζεται περισσότερο και πιο αποτελεσματικά γίνονται ασκήσεις εικονικές, οι οποίες όμως ποτέ δεν μπορούν να δοκιμάσουν ε, στην πράξη την αποτελεσματικότητα του συντονισμού, όπως δυστυχώς οι πραγματικές θεομηνίες. Στην παρούσα κρίση, χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούν το MIC για να δουν πώς μπορούν να βοηθήσουν και να χρησιμοποιήσουν τις δικές μας διευκολύνσεις για να χορηγήσουν ανθρωπιστική βοήθεια. Τρίτον, δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι στη δεύτερη επιτροπή του ε, Μπαρόσο η ανθρωπιστική βοήθεια και η πολιτική προστασία είναι στο ίδιο χαρτοφυλάκιο και είναι πολύ σημαντικό πραγματικά στοιχείο. Επιπλέον, τώρα έχουμε και η πάτη εκπρόσωπο με διπλή ιδιότητα και θα έρθω συνέχεια σε αυτό, δεν είναι μόνο στο εσωτερικό της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά είναι και ζήτημα των κρατών μελών, αλλά και του Συμβουλίου. Οπότε η όλη ιδέα της διπλής ιδιότητας που κρύβεται πίσω από την ύπατη εκπρόσωπο είναι ακριβώς αυτό. Να συνεργάζονται καλύτερα και να συντονίζονται καλύτερα Συμβούλιο και Επιτροπή. Και φάνηκε και από την κρίση αυτή ότι ήταν πρόοδος η αλλαγή αυτή. Τέλος, θα ήθελα επίσης να πω το εξής. Με έχουν στεναχωρήσει λίγο κάποιες ε, παρατηρήσεις. Βέβαια, ως Επίτροπος δεν μπορεί να στεναχωριέμαι, σημειώνω απλώς αυτά που λέτε. Αλλά ε, όλοι όσοι εργάζονται από την πρώτη ώρα επιτόπου μερά νύχτα στις Βρυξέλλες και το Σαββατοκύριακο χωρίς να παραπονούνται, χωρίς να ζητούν υπερορίες και αποζημίωση εργάζονται πάρα πολύ σκληρά και μέσα σε λίγες ώρες επιτόπου είχαμε παρουσία και βοήθεια παρόλο που εκεί οι δυνατότητες και τα μέσα τους ε, επλήγησαν σφοδρότατα, σφοδρότατα. Λοιπόν, σας παρακαλώ, καταλάβετε ότι πρόκειται για μαζική καταστροφή, απρόβλεπτη, και μπορεί κανείς να απαντήσει μόνο εφόσον συμβεί και να αποδείξει ότι μπορεί να οργανώνεται σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι το έχει αποδείξει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη μαζικά και άμεσα επίσης ε, υποστήριξαν τη δράση αυτή και ας κάνουμε λίγο, ε, λιγότερη κριτική στις υπηρεσίες μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η συζήτηση έληξε η ψηφοφορία επί του σχετικού ψηφίσματος θα διεξανθεί κατά την περίοδο της ε, Συνόδου του Φεβρουαρίου, της πρώτης. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η δήλωση της ΥΠΑ εκπροσώπου της Ένωσης για τις εξωτερικές υποθέσεις και την πολιτική ασφάλειας και αντιπροέδρου τη Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση στο Ιράν. Πάμε αρκετά γρήγορα. Όπως βλέπετε δεν έχετε χρόνο για να μπορέσετε